Δηλαδή ε, θα πρέπει ε, η Ευρώπη είτε να εφαρμόζει τα συμμεφωνημένα αλλά εν πάση περιπτώσει διαφορετικά να ε, επιζητήσει άλλες λύσεις. Ευχαριστώ. Έληξε η συζήτηση και το αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Meine sehr Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι η έκθεση του κυρίου Κάζα σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας και διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατωτάτου κανονικού συντελεστή. Θα συνεχιστεί η συζήτηση. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο εισηγητής κύριος Κάζα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι σημαντική η ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Έχει καθυστερήσει αυτή η ψηφοφορία και γι' αυτό απουσιάζουν πολλά από τα μέλη. Μόλις ε, ξεκίνησε. Όπως λοιπόν σωστά δήλωσε και η Πρόεδρος, η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική διότι αφορά το θέμα του ΦΠΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας και τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Όπως ξέρετε, οι διαπραγματεύσει για τη διόρθωση του συστήματος και για την ε, υιοθέτηση ενός σταθερού συντελεστή είναι μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και καιρό. Το μεταβατικό σύστημα που έχει αρχίσει να ισχύει από το 1993 έχει παραταθεί επαριλημμένος. Και όπως ξέρουμε, η κατάσταση ως έχει δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ε, πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη, σταθερή λύση. Το μεταβατικό σύστημα που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή δεν δίνει τα ε, επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά. Δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι αποτελεσματικές. Επίσης, παρακολεί την αποτελεσματικότητα των διακρατικών συναλλαγών των επιχειρήσεων. Έτσι, το σύστημα αυτό γίνεται ευάλωτο σε πολύπλοκες ε, μορφές απάτης, όπως η κυκλική απάτη, η απάτη καρουζέλ, κάτι που το έχουμε συζητήσει και πρόσφατα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες και για το εισόδημα που εισπράττουν τελικά τα κρατημέλη. Η λύση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι απλή. Πρέπει να, ε, να ζητήσουμε μία ικανοποιητική λύση, αλλά αυτό θα γίνει μόνο μετά από μια διεξοδική συζήτηση και μια καλή οργάνωση γύρω διαβουλεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα μα καθησύχασε ότι θα δημοσιεύσει μια πράσινη βιβλό ώστε να συζητηθεί το, σύστημα, το θέμα αυτό. Η έκθεση της οποίας αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει τη σύνταξη θέλει να καλέσει την Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι η προσέγγιση θα είναι αποτελεσματική και ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε ένα νέο σύστημα που θα κάνει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική. Κατά δεύτερον, το νέο αυτό σύστημα θα πρέπει να άρει το άχθος ε, για τον τομέα των επιχειρήσεων σε, μεγάλο, σε μεγαλύτερο βαθμό και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά και την απάτη. Η έκθεση αυτή, όπως τα ξέρετε, ήδη υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και καλή παροτρύνει την Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι θα δημοσιευτούν χειροπιαστέ προτάσεις ω το 2013. Το τονίζω αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα υιοθετηθεί και θα αρχίσει να ισχύει από το 2013 απλώς, αλλά θα πρέπει προτάσεις να δημοσιευτούν τουλάχιστον το 2013. Άρα, εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε στην ανταλλαγή απόψεων, στον εντατικό διάλογο, στο το σύστημα να θεσπίσει, να αρχίσει να ισχύει πριν από την εκπνοή του μεταβατικού συστήματος. Να μην χρειαστεί να παραταθεί κι άλλο το μεταβατικό αυτό σύστημα. Για την, ανανέωση, για την υιοθέτηση λοιπόν του νέου συστήματος ελπίζουμε ότι θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις που θα βασιστούν και σε καινοτόμε λύσεις. Να ευχαριστήσω λοιπόν εδώ όλους τους συναδέλφους και τους σκιώδει εισηγητέ και να πω ότι ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση για το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάζα. Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο επίτροπο Μέτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως τον κύριο Κάζα για την ε, επικοδομητική έκθεση ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνουμε κατά πέντε χρόνια το ποσοστό του ΦΠΑ. Η ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επιτρέψει να προχωρήσει πρόταση πριν από το τέλος του έτους προτού τελειώσει η τρέχουσα ισχύς της της ε, ε, ρυθμίσεως. Δεν φαίνεται να υπάρχει δυσκολία και όπως είπε και ο Ντέβιτ Κάζα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας επιτρέψει να έχουμε νομική βεβαιότητα και να προωθήσουμε το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σκεφτεί το μέλλον του ΦΠΑ για να αξιολογήσει τις διάφορες ατέλειες του συστήματος, το πολύπλοκο χαρακτήρα, ε, το βάρος ε, των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ούτω καθεξής. Πριν από το τέλος του, του έτους θα προτείνω να ε, δημοσιεύσουμε μία πράσινη βίβλο για την ολοκλήρωση του συστήματος και την καλύτερη πρόταση για το μέλλον. Προσβλέπω στις αντιδράσεις σας για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μία, ένα πιο απλό σύστημα και πώς θα μειώσουμε το κόστος για τις ε, επιχειρήσεις ε, συγχρόνως μειώνοντας ε, την διαφθορά και βελτιώνοντας την κατάσταση στα κλάτη μελη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατυπώσει την πολιτική της στο ΦΠΑ και να διατυπώσει μια πρόταση που να ισχύσει από το τέλος του 2011. Αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής του ΦΠΑ και προσβλέπω σε έναν επικοδομητικό διάλογο μαζί σας αργότερα. Αλλά οι τροπολογίες αυτές είναι εκτός της εμβέλειας της προτάσεως που συζητάτε σήμερα όπου μιλάμε ε, για τις περιοδικές ανανεώσεις ή επεκτάσεις. Οι ε, ρυθμίσεις ε, οι νέες θα γίνουν βαση της πράσινης βίβλου και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσει μέχρι το 2013 ένα νέο έγγραφο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεσμευτούμε πότε θα διατυπώσουμε μια σαφή πρόταση για το ποσοστό του ΦΠΑ και ε, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή πιο ευρέως. Ελπίζω όμως ότι η διαβούλευση αυτή θα δώσει ε, μια σαφή ιδέα για τις προτεραιότητες του ΦΠΑ και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξαρτηθούν από αυτή τη διαβούλευση και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στους ε, αγορητάς των πολιτικών ομάδων για το Λαϊκό Κόμμα τώρα για ένα λεπτό και μισό έχει το λόγο η κυρία Εσέγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επικεντρώνεται στην συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος ως το 2015. Οπότε και θα έχουμε ε, μια περικοπή κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ούτως ώστε να μην έχουμε ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού και ε, αυτό το οποίο εμείς κυρίως πρεσβεύουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανέλθει με νέα φάση διαβούλευσης όσον αφορά την θέσπιση ενός συστήματος ΦΠΑ. Ορισμένες δε εκ των προτάσεων που έχουμε υποβάλει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί δείχνουν την ορότα που θέλουμε να ακολουθήσουμε όσον αφορά το ΦΠΑ για να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του ΦΠΑ για να διευκολύνουμε τις ΜΜΕ και επίσης να αποφύγουμε τις ε, σχετικές φορολογικές παραβάσεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα σε πολλά κράτη-μέλη και ένα από τα προβλήματα είναι το τι θα γίνει με τον ΦΠΑ, εάν θα αυξηθεί και εάν θα βοηθήσει. Πάντως εκεί όπου βασιλεύει η απάτη δεν θα ωφελήσει η αύξηση του συνδυαστή ΦΠΑ. Πρέπει να καταπολεμηθεί πρώτα πρώτα η απάτη και θέλουμε μια σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και για δύο λεπτά Ζητεί το λόγο ο κύριος Κούτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. A Consiliului, cota minimă a TVA a asigurat funcționarea sistemului la un nivel acceptat. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ο ΦΠΑ ε, λειτουργεί σωστά αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμπεράσματα από τις διάφορες κρίσεις στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον ε, ε, ΦΠΑ για να καταργηθούν τα εμπόδια τα οποία ακόμη μας εμποδίζουν. Θα πρέπει επίσης να προβούμε και στην καταπολέμηση της της ε, διαφθοράς και πιστεύω ότι ε, αν, ε, αν επεκτείνουμε το ισχύον σύστημα μέχρι το 2015 θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε το σχετικό περιβάλλον και να έχουμε καλύτερες προπτικές για κατάρτιση ενός καλύτερου συστήματος. Υπάρχουν όμως ορισμένες κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν να αυξήσουν το ΦΠΑ στο 24%. Παραδείγματος χάρη στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Μέχρι στιγμής οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει να διατηρήσουν το ΦΠΑ σε επίπεδο 10% αλλά ε, εάν ε, υπάρξει υπέρβαση αυτού του περιθωρίου θα χρειαστούμε ε, νέα, νέα νομοθεσία και θα πρέπει πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, οι λαοί ε, ε, υφίστανται μία κατάσταση φτώχειας και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να ληφθεί υπόψη και το εισόδημά τους. Κύριε Κούτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα για τους φιλελευθέρους έχει το, δίκιο, το λόγο συγγνώμη, για 1,5 λεπτό ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τον εισηγητή διότι θα πρέπει να αποφύγουμε την τυθάσευση του πληθωρισμού με μεταβολή των συνδυαστών του ΦΠΑ διότι έτσι παραβλάπτουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της ελευθέρας ε, αγοράς και πάρα πολύ σωστά ο εισηγητής όσον αφορά την ε, ενιαία αγορά ότι ακόμα και σήμερα οι ρυθμίσεις μπορούν να επιδράσουν αρνητικά. Γι' αυτό και εμείς ζητούμε ένα καθορισμένο, πάγιο σύστημα ε, συντελεστές που να ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα προσθέσουμε την ελεύθερη ενιαία αγορά. Έτσι θα εξυπηρετήσουμε και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί η γραφειοκρατία σχετική με την υποβολή του ΦΠΑ και επίσης ε, να δούμε πώς θα έχουμε φορολογική πολιτική που θα βοηθά, δεν θα παρεμποδίζει τις ε, ΜΜΕ. Ταυτόχρονα θα δομήσουμε και την απάτη. Ε, Βεβαίω, είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας η φορολογική πολιτική, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι μια ενιαία αγορά απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία, ακόμα και στα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Θα πρέπει επομένω να τολμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα στην επόμενη πρότασή τη και επομένω να καταλάβει ότι σωστή αφετηρία είναι η θέσπιση σωστών μέτρων για το ΦΠΑ. Δύσκολη είναι η καιρή και χρειάζονται επομένω προσεκτική ανάλυση οι κινήσει μα. Ευχαριστούμε κύριε Σνίτλε, ο πρόεδρο. Και τώρα έχουμε την ώρα του Catch the Eye. Κυρία Μπασέσκου, ένα λεπτό. Α, που απουσιάζει η κυρία Μπασέσκου. Καλά. Κάτι διάει, αλλά το μάτι δεν τη βλέπει. Και για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, μέλη της Επιτροπής. Η προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ε, ένα ε, σύστημα μέχρι το 2015. Καταλαβαίνω τον ε, στόχο που είναι να υπάρξει μία ενιαία κατάσταση αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τίνουμε σε μία μεγαλύτερη εναρμόνιση διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου διαπιστώνουμε ότι το σύστημα του ΦΠΑ είναι πολύ κακά οργανωμένο στην Ευρώπη και επίσης είναι κακά οργανωμένοι και οι κανόνες οι οποίοι διέπουν τα εθνικά, το εθνικό εμπόριο, το εμπόριο σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις επιτρέπεται η φοροδιαφυγή να έχει σχεδόν νόμιμη μορφή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεών μας το σύστημα του ΦΠΑ να εξεταστεί και να επαληθευτεί. Θεωρώ ότι το 2013 είναι ρεαλιστική ημερομηνία και το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να επιληθεί με καλύτερους κανόνες. Για να δευτώ κύριος Μπρόνς. Κύριε Μπρόνς. Το αναγκαίο κακό πάντοτε σχετίζεται και με τις ανάγκες για τις δαπάνες. Όμως η φορολογική πολιτική για το πώ θα λάβουμε τα χρήματα των φορολογουμένων είναι κάτι που είναι σημαντικό να έχει καθοριστεί από πριν για το να καταλήξουμε σε έναν κοινό σταθερό συντελεστή, κάτι που είχε προγραμματίσει η Επιτροπή το 1993, θα πάρει τις εξουσίες από τα χέρια των κρατών μελών. Θα έχουν πλέον ε, χάσει και σε αυτό το θέμα την κυριαρχία του στα κράτη-μέλη και θα είναι ουσιαστικά χωρίς δύναμη τα κράτη-μέλη μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει αναλάβει την κοινή φορολογική πολιτική. Η πολιτική λοιπόν ως τώρα ε, είναι για ενοποίηση του συστήματος και για εδραίωσή του, όχι για να χάσουν τις κουσίες του τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς. Κυρία Μπασέσκου, εφόσον Επιστρέψατε, σας δίνουμε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά βρισκόμουν σε άλλη συνεδρίαση. Η νέα στρατηγική για τον ε, φόρο προστιθέμενη αξία θα πρέπει να περιορίσει το διοικητικό άχθο για τι επιχειρήσει καθώ και τα φορολογικά εμπόδια. Θα πρέπει να βελτιώσει το χώρο των επιχειρήσεων, των συναλλαγών των εμπορικών, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, θα πρέπει λοιπόν για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσει αυτέ να μην, να μην βρίσκονται πλέον σε μειονεκτική θέση, όπω τώρα συμβαίνει. Το σημερινό σύστημα ΦΠΑ δεν επιτρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή, να αναλύσει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή τη και να διαβουλευθεί με ειδικού ώστε να καθορίσει μια νέα στρατηγική για το φόρο προστιθέμενης αξία, που να είναι ωφέλιμη και ε, μάλλον υποφελή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν οι φόροι να περιοριστούν ώστε να μην μειώνουν τι δυνατότητε ε, συλλογή εισοδήματο και βεβαίω να καθοριστεί πολύ συγκεκριμένα και ο το, ο τόπο συλλογή του φόρου για τις ενδοκινοτικές συναλλαγέ. Ευχαριστούμε τον λόγο τώρα ο επίτροπο. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις ιδέες σα, αυτή τη συζήτηση. Με ικανοποίηση διαπιστωρώ ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν κοινέ ιδέε για την ανανέωση του ισχύοντος συστήματο ΦΠΑ. όπω είπα και στις αναρτήριε παρατηρήσει μου, οι τροποποιήσεις, οι διορθώσει του συστήματο έχουν άμεση σχέση με το μέλλον τη φορολογική μα πολιτική και το ΦΠΑ. Η Επιτροπή λοιπόν ξέρει ότι η τεχνική αυτή πρόταση έχει να κάνει μόνο με την προσωρινή παράταση των ελάχιστων προδιαγραφών για τον συντελεστή ΦΠΑ. Όμως, το το αποτέλεσμα των ε, διαβουλεύσεων για μια νέα στρατηγική του ΦΠΑ είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι πρόημο αυτή τη στιγμή βεβαίω να ορίσουμε ένα κοινό επίπεδο κατώτατου συντελεστή. Ένα κατώτατο επίπεδο μάλλον κοινού συντελεστή. Όμω θα πρέπει να έχουμε υπόψη του στόχου και το πλαίσιο τη νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ και το πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ω τώρα. Να επαναλάβω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεσμευτεί ήδη σήμερα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία για τη μελλοντική νομοθετική τη πρόταση για του ε, συντελεστέ. Θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ενδελεχώ για το μέλλον του ΦΠΑ και να έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποιε είναι οι προτεραιότητε τη Επιτροπή σε μια πρώτη φάση. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών θα καθοδηγήσει το μελλοντική πολιτική τη Επιτροπή για την νομοθετική πρόταση για το ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή περατώνουμε το έργο μα ε, για το θέμα αυτό και όπω ξέρετε τι ερχόμενε εβδομάδε θα έχουμε τον πραγματικό διάλογο, τις ερωταπαντήσεις για το θέμα αυτό και με το κοινό συζήτηση θα γίνει και με τα μέλη του Κοινοβουλίου και με τους εκπροσώπους των κρατών μελών Είναι σαφέ λοιπόν ότι τα ζητήματα που σήμερα αναφέρθηκαν θα τεθούν σε αυτέ τι συζητήσει. Ε, ελπίζω λοιπόν να έχουμε συζητήσει πραγματικά επικοδομητικέ του ερχόμενου μήνε και αφήστε λίγο χρόνο στην Επιτροπή ώστε να καταρτήσει μια πολύ ε, ε, πιο εύρωστη πολιτική ΦΠΑ για το προ ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο, κύριο Σκάζα. Έχετε το λόγο. Eh, Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μεταφράζεται ο μιλητή. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Τώρα αποκαταστάθηκε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως προείπαμε θα πρέπει να καταπολεμηθεί κάθε φαινόμενο απάτης. Παντού στο σύστημα του φόρου προσθεμένης αξίας θα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις ε, και να αρθούν όλοι οι φραγμοί στην ε, ακόλυτη δραστηριότητά τους όπως ε, έχει σήμερα η κατάσταση και έτσι να είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία τους και της ενιαίας αγοράς επίσης δεν επισήλθαμε στις λεπτομέρειες όσον αφορά τις προτινόμενες λύσεις αλλά αυτό το οποίο ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να συζητηθεί επαρκώς το καινούργιο σύστημα. Πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό το νέο σύστημα από ότι το ισχύον. Αυτός είναι ο στόχος της ε, έκθεσης μου. Εκεί θέλω να επισύρω την προσοχή της. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς κάποιες προτάσεις της. Και με αυτές τις προτάσεις να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο δίκαιο σύστημα ΦΠΑ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσα. Στις 11.30 αύριο θα γίνει ψηφορία αυτής της έκθεσης και τώρα. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Βοήθεια κατεπίγουσα προς την IT. Η κυρία